θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι οι προφορικές ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αναθεώρηση του μονίμου πλαισίου για την κράτηση στοιχείων. Ο κύριος Σαλβάρο είναι ο πρώτος που έχει το λόγο. Herzlichen Dank, Herr σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, με κύριε και κύριοι. Δεν είναι η πρώτη φορά που συζητούμε το θέμα αυτό. Είναι η πρώτη φορά ίσως αυτή την ώρα της ημέρας, αλλά το ερώτημα γεννάται σιγά σιγά πότε πλέον θα ολοκληρωθεί η συζήτηση στο θέμα αυτό της διακράτησης προσωπικών δεδομένων. Είναι πολλά τα δικαστήρια, συνταγματικά, ε, συνταγματικά κυρίως δικαστήρια, τα οποία έχουν κρίνει πως είναι αντισυνταγματική η διακράτηση αυτών των στοιχείων. Το Ιρλανδικό Συνταγματικό ε, δικαστήριο μαζί με προδικαστικό ερώτημα προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αλλά και πολλοί άριθμα κράτη-μέλη εκδηλώνουν όχι μόνο τη δυσφορία τους, την αδυναμία να κατανοήσουν αλλά και την απόλυτη απόρριψη αυτών των ε, θέσεων περί διακράτησης προσωπικών δεδομένων. Λυπούμε διότι πριν από τέσσερα χρόνια ήδη είχαμε κάνει διαπιστώσεις που αποδεικνύονται σωστές. Από το 2005 ουσιαστικά και έχουμε και από νομομαθείς και από, και από θέματα τεχνικού χαρακτήρα και για λόγους κοινωνικούς επίσης έχουμε απορρίψει αυτή τη διακράτηση προσωπικών δεδομένων και αποδεικνύεται ότι ήμασταν σε κάθε επίπεδο ε, εύστοχοι στις παρατηρήσεις μας, επισημάνσεις μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως επιμένει και από την ε, Επιτροπή περιμένουμε να δώσει, να δώσει απαντήσεις ως προς το πώς θα χρησιμοποιούνται από τις ε, αρχές ε, της αστυνόμευσης, από τις κρατικές αρχές, τα στοιχεία αυτά. Δεν αποδεικνύεται πουθενά κατά πόσον είναι απαραίτητα τα στοιχεία αυτά. Και γι' αυτό πολύ σωστά διατυπώνεται το ερώτημα του πότε θα γίνει ή πότε μπορούμε να περιμένουμε την κωδικοποίηση, την νομοθετική δηλαδή διατύπωση αυτών των θεμάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αυτή τη θητεία ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πρόταση νομοθετική και κυρίως ιδιαίτερος να δούμε τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό. Ελπίζω έστω σήμερα το βράδυ να ενημερωθούμε, να ακούσουμε λίγο περισσότερα πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, Μπορείτε να με ενημερώσετε, γιατί βλέπω αστεράκια πάνω στον ε, πίνακα. Μπορείτε να με ενημερώσετε αν έχω ξεπεράσει το χρόνο ομιλία μου ή έχει γίνει κάποιο σφάλμα, γιατί νόμιζα ότι είχα περισσότερο χρόνο. Πώ ε, είναι δυνατόν να καλύψουμε λοιπόν το θέμα αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε διεξοδικά το θέμα και να καταλήξουμε στι τελικέ αποφάσει. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για αυτή την εισαγωγή που κάνατε. Πραγματικά επρόκειτο περί εισαγωγής και ζητώ από τους επόμενους αγορητές να τηρήσουν παρακαλώ το χρόνο που τους διατίθεται. Η κυρία Σατζεντίνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Οι πράσινοι έχουν μια πολύ απλή ερώτηση για την Επίτροπο. Πότε αναμένεται να έχουμε την αναθεώρηση το πλαίσιο για τη διακράτηση των στοιχείων που ισχύει. Μπορείτε να απαντήσετε πολύ γρήγορα, ε, κυρία Σατζεντίνη, στην κυρία διότι περίμενε επιμακρών την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Αλλά φοβούμαι ότι δεν είναι η απάντηση επιθυμητή που θα μας δώσετε. Φαίνεται ότι έχετε αμελήσει την αναθεώρηση ε, του πλαισίου για τη διακράτηση των στοιχείων. Γιατί τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι είναι χρήσιμο το πλαίσιο αυτό διακράτηση των στοιχείων. Όμως, χρειαζόμαστε να έχουμε ένα κάποιο πλαίσιο ούτω ώστε να προστατεύεται η ιδιωτική ζωή ε, των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό το πλαίσιο όμως ε, παραβιάζει τα δικαιώματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής των πολιτών, συλλέγει και ε, κρατά στοιχεία για τους Ευρωπαίους πολίτες, δεν έχει αναθεωρηθεί το πλαίσιο για τη διακράτηση των στοιχείων και πρέπει να κάνετε κάτι για το όλο πρόβλημα. Κανείς δεν επιβεβαιώνει ότι λειτουργεί αυτή η οδηγία. Αν δεν λειτουργεί η οδηγία, ας απαλλαγούμε από την οδηγία και ας βρούμε εναλλακτική λύση. Ας πούμε ένα σύντομο πάγωμα ε, όπου χρησιμοποιούμε την νομοθεσία, τους ε, εμπειρογνώμονες συλλέγονται τα στοιχεία από την αναγκαία, διατηρούνται μόνο όσο είναι αναγκαία όταν υπάρχουν υπόνοιες για κάποιον Λοιπόν, κυρία Επίτροπε, μπορείτε σας παρακαλώ να δώσετε μια απάντηση στα κράτη-μέλη γι' αυτό. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις που υπάρχουν ερωτηματικά. Πολλοί πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν να προστατεύσουν την ιδιωτική του ζωή και θέλουν να σας βοηθήσουν να αντικαταστήσετε αυτή την οδηγία με κάτι που είναι πολύ καλύτερο. Η κυρία Διόμ είναι η επόμενη. Κυρία Επίτροπε, συνάδελφοι, Χαίρομαι που γίνεται λόγο η, οδηγία η συζήτηση για την ανθεώση οδηγία του 2006, έστω και καθυστερημένα. Πρόκειται για μια συζήτηση που πρέπει να γίνει. Και τη χρειαζόμαστε. Και τη χρειάζονται και οι πολίτες που αναρωτιούνται όλο και περισσότερα, περισσότερο για το ποια είναι η τύχη των προσωπικών τους δεδομένων. Η οδηγία αυτή είναι επίμαχη σε πολλά σημεία. Αυτό φαίνεται από, τις, την ακύρωση της μεταγραφής τους, της μεταγραφής της οδηγίας σε διάφορες περιπτώσεις όπως στη Ρουμανία, τη Τσεχία και τη Γερμανία. Η οδηγία ε, παρεμβαίνει στην προσωπική ζωή ε, ασφαλώς και δεν τίθεται θέμα για διατήρηση στοιχείων που συνδέονται με κάποια ποινική δίωξη. Ε, όμως εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα για, τις, για το άλλου τύπου περιπτώσεις. Θα ήθελα να μας δώσετε απαντήσεις ανάλογες με τις ανησυχίες μας σε πολλά σημεία. Για παράδειγμα, το ότι πρέπει να αποδεικνύεται η ανάγκη και η αναλογικότητα μιας τέτοιας, ενός τέτοιου μέτρου και επίσης να καλύπτεται συγκεκριμένος στόχος, ε, κάτι το οποίο ερμηνεύεται διασταλτικά από τα κράτη-μέλη και το πώς η συντήρηση, η διατήρηση των στοιχείων μπορεί να γίνει με τρόπο που να παρεμβαίνει λιγότερο στην ιδιωτική σφαίρα των ανθρώπων. Σε μια κοινωνία όπου η τεχνολογία της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών είναι πανταχού παρούσες, η, τα, η, η προστασία των προσωπικών στοιχείων ε, είναι απαραίτητο να γίνεται με πιο αυστηρό τρόπο, να μην είναι μόνο θεωρητική. Ευχαριστώ. Thank you very much. And... ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ernst την επόμενη. Ευχαριστώ πολύ. Μια ατέρμονη ιστορία, δεν ξέρω ούτε πόσες φορές την έχουμε συζητήσει. Και είναι ένδειξη παινίας νομίζω το ότι χρειάζεται να καταθέσουμε προφορική ερώτηση για να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι σκοπεύει να κάνει για το θέμα αυτό. Αντί λοιπόν να αποδεχόμαστε τα τετελεσμένα, καλό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανοίξει τα χαρτιά της και να μας πει τι σκοπεύει να κάνει. Ούτως ή άλλως συμφωνία για την αποθήκευση έχει αποτύχει. Ο στόχος της προστασίας των προσωπικών δεδομένων δεν έχει επιτευχθεί. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία λόγω των αποφάσεων των σταγματικών δικαστηρίων δεν είναι σε θέση να εφαρμόσουν την οδηγία, ενώ κάποια άλλα, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να χρειαστούν έξι, μπορεί να, κρατάνε, τα στοιχεία έξι μήνες, άλλα δώδεκα, άλλα για πιο σημαντικά εγκλήματα, άλλα για λιγότερο σημαντικά δικήματα. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με ένα μοσαϊκό διαφορετικών νομοθεσιών που επηρεάζει αρνητικά και την εσωτερική αγορά και πάντως δεν διευκολύνει τις αστυνομικές αρχές στην δίωξη του εγκλήματος από ό,τι μας λέει τουλάχιστον η γερμανική αστυνομία. Ερωτώ λοιπόν από πού αντλείται αυτή τη ε, βεβαιότητα και τη στάση που τηρείται. Υπάρχουν τόσες αναλύσεις της κατάστασης ε, από τις ε, υπηρεσίες της γερμανικής αστυνομίας του 2011, επί παραδείγματι, που μας λένε ότι δεν μπορεί να προκύψουν χρήσιμα δεδομένα από την αποθήκευση αυτών των στοιχείων ή από το Ινστιτούτο Max Planck, μελέτη του 2012, μας λέει ότι δολοφονίες, παιδική πορνογραφία, ε, ε, εγκληματικότητα μέσα από το διαδίκτυο, ληστείες δεν καλύπτονται από αυτά τα διακρατούμενα δεδομένα. Ερωτώ λοιπόν κυρία Μάλιστρου, αν πρόκειται να κάνετε τη δουλειά σωστά ως Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να προχωρήσετε ε, να επιμείνετε στην εφαρμογή της οδηγίας μέχρι να εκδοθεί σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και να αναθεωρήσετε τότε τις θέσεις σας και την νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ και ο επόμενο ομιλητής είναι ο κύριος Φως. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η 15χρονη Αμάντα Τότ από τον Καναδά και η τύχη της μας απέδειξε για άλλη μία φορά ότι μπορεί να κυκλοφορήσουν εις βάρος ενός παιδιού μέσα από το ίντερνετ, από το ίντερνετ ε, στοιχεία που μπορούν να κάνουν τεράστιο κακό. Το ο διασυρμός μέσα από το ίντερνετ δεν μπορεί να, αντιμετωπιστεί μέσα από τα συστήματα αυτά. Η παιδική πορνογραφία, η εγκληματικότητα μέσα από το ίντερνετ ή και το λεγόμενο απλό phishing επίσης δεν αντιμετωπίζονται Το ΔΕ Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση των ναρκωτικών έχει μιλήσει και για το θέμα αυτό της κατακράτησης δεδομένων. Βεβαίως χρειάζεται μια ισορροπημένη, ένα ισορροπημένο μείγμα μεταξύ της διακράτησης δεδομένων αλλά και μιας δικαστικά, υποδικαστική εποπτεία προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η υπόθεση της μικρής Αμάντα Τότ δείχνει ότι οι ανώνυμοι χρήστες του διαδικτύου μπορούν να είναι υπέτοιοι για πολύ σοβαρά εγκλήματα εφόσον έχουν τη δυνατότητα της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα. Δεν υπάρχει όμως λύση. Τη λύση δεν μας τη δίνει η διακράτηση προσωπικών δεδομένων και επιτυχίες των διοκτικών αρχών, όπως στην περίπτωση του ε, τρομοκράτη της Τουλούζ, της Τουλούζης μας δείχνουν ότι μπορεί να είναι σε ορισμένες περιπτώσεις χρήσιμα τα δεδομένα, ωστόσο η οδηγία στην τωρινή της μορφή δεν φαίνεται να έχει εξασφαλίσει επαρκή ισορροπία και ως εκ τούτου φαίνεται πολύ πολύ σημαντικό να προκύψουν νέες προτάσεις και επί τη βάση των αξιολογήσεων του 2011 νέα και καλύτερη πρόταση για συζήτηση. Πέραν αυτού και ανεξαρτήτως αυτού είναι απαράδεκτο το ευρωπαϊκό δίκαιο και η τήρησή του να είναι να τίθεται να αμφιβόλο από τη ίδια τη Γερμανίδα της ε, Υπουργό της Δικαιοσύνης. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα εκπρόσωπος του Υπουργείου ε, Δικαιοσύνης της Γερμανίας σε μια συνεδρίαση της Επιτροπής των Αναφορών μας είπε ότι η γερμανική κυβέρνηση σκοπεύει να μην καταθέσει πρόταση ως προς την οδηγία για τη διακράτηση προσωπικών δεδομένων. Και όσο η μεταφορά ε, σε ε, εθνικό επίπεδο και η εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας δεν έχει προχωρήσει, δεν θα προσφερθούν στοιχεία από πλευράς της Γερμανίας. Επομένως, ερωτώ τι είδους χρησιμότητα μπορεί να έχουν αυτά τα στοιχεία. Άλλωστε και εσείς, κύριε Επίτροπε, έχετε πει, έχετε δηλώσει στην ε, διαδικασία που εγώ έχω, κινήσει, έχω ζητήσει να κινηθεί επί παραβάση των συνθήκων κατά της Γερμανίας, ότι δεν μπορείτε να αντιδράσετε σε αυτή την άρνηση των γερμανικών αρχών. Άρνηση να προσφέρουν στοιχεία που διακρατούν. Κάθε κράτος μέλος είναι υποχρεωμένο να εφαρμόζει ουσιαστικά το ευρωπαϊκό δίκαιο και μέσα στις προθεσμίες, όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Έτσι λοιπόν η Γερμανίδα Υπουργό Δικαιοσύνη μα λέγει ότι δεν είναι δυνατόν να υλοποιήσει μέσα στι προθεσμίε την οδηγία. Αυτό είναι απαράδεκτο. σω λοιπόν είστε σε θέση να προσφέρετε με την τοποθέτηση σα κάποιε ε, προτάσει. Αλλά νομίζω και η Αυστρία έχει αρνηθεί να υλοποιήσει την ε, οδηγία και, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να βρούμε μία λύση η οποία θα είναι και σταγματικά αποδεκτή και πρακτικά εφαρμόσιμη. Ευχαριστώ πολύ. Μπλε κάρτα από τον κύριο Αλβάρο. Δέχεστε. Κύριε Φω, να απαντήσετε στην ερώτηση του κύριου Αλβάρο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φω, ε, για το όσο είπατε. ακριβώ για το για την Υπουργό Δικαιοσύνης. Δεν θεωρείτε ότι η Υπουργός Δικαιοσύνης έχει καθήκον εφόσον ε, εντοπίζει ότι κάποια διάταξη μπορεί να είναι αντίθετη με το δίκαιο και προκειμένου πρόκειται για ζήτημα συνταγματικό. Δεν θα πρέπει η υπουργό αυτή να αναλάβει την πρωτοβουλία και ιδιαίτερα αν κινδυνεύει γενικότερα και το ευρωπαϊκό δίκαιο, όχι μόνο το σταματικό, να δηλώσει ότι μέχρι ότου υλοποιηθεί κάτι το πιο ε, αποδεκτό να ε, αναβάλει την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας. Ευχαριστώ κύριε Φως, θα δεχθείτε άλλη μια μπλε κάρτα από την κυρία Νετφέλτ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Νετφέλτ. Ε, Με έκπληξη ακούω τον συνάδελφο τον κύριο Φως να αναφέρεται στο παράδειγμα της Τουλούζης ε, ε ως επιτυχία των αρχών. Ε, ήταν μια καταστροφή. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν γνωστός στις μυστικές υπηρεσίες ε, που ήταν στο κατάλογο των ε, επιβατών που αρνούνταν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα αεροπλάνα τους που ε, ήταν, είχε πάει στο Αφγανιστάν το ξέραμε και, αυτόν τον αφήσαμε και ξανασκότωσε λοιπόν ποια είναι η επιτυχία πραγματικά δεν καταλαβαίνω Mr. Foss για το θέμα το σχετικό, την ερώτηση σχετική με την Υπουργό Δικαιοσύνη. Κοιτάξτε, δεν έχει πει το Γερμανικό Σταγματικό Δικαστήριο ότι η οδηγία αυτή είναι ε, αντισταγματική. Έχει πει ότι ή έχει επισημάνει ότι ο νόμος περί εισαγωγής στο εθνικό δίκαιο της εν λόγω οδηγίας δεν επιτρέπει επαρκέ επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων, δηλαδή σε εθνικό επίπεδο προστασία των δεδομένων είναι πολύ χαμηλή. Αυτός είναι, αυτό είναι το, αυτή είναι η αιτιολογία πάνω στην οποία στηρίζει την απόφασή του το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο και ως εκ τούτου θα πρέπει οι δεσμεύσει τι οποίε έχουμε αναλάβει σε ευρωπαϊκό επίπεδο εμεί να τι υλοποιήσουμε ουσιαστικά στη Γερμανία. Για την άλλη ερώτηση, για την Τουλούζη πάντοτε πρέπει να λέμε ότι χρειάζονται αποδείξεις, απτές αποδείξεις που μπορούν να οδηγήσουν σε καταδίκη, σε δικαστήριο. Μόνο έτσι μπορούμε να αξιοποιήσουμε ουσιαστικά τα ε, προσωπικά αυτά δεδομένα. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Επίτροπο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που γίνεται η συζήτηση και εγώ. Θα μου δώσετε έτσι την ευκαιρία να διευκρινίσω κάποια πράγματα και να σας εξηγήσω και τις προθέσεις μας. Η Κομισιόν, όπως έχει ανακοινωθεί επανειλημμένως και στην ε, ε, αξιολόγηση έχει σκοπό να ε, προτείνει να κάνει κοινέ προτάσει. Η Κομισιόν είχε κάνει την αρχή τη πρόταση το 2005, αλλά αναγνωρίζει ότι τα δεδομένα τηλεπικοινωνιών ε, χρησιμοποιούνται πολύ και διατηρούνται ε, σε ποινικέ διώξει για πολύ σοβαρά εγκλήματα. Συνεπώ, είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούνται αυτά τα στοιχεία από τη δικαιοσύνη. Ήταν και παραμένει απαραίτητο να εγγυηθούμε ότι μέσα στα πλαίσια της αναλογικότητας και με συγκεκριμένες ε, μέτρα ασφαλείας τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να, είναι, να διατίθενται ε, για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα αν τα χρειάζεται η αστυνομία. Οι διαδικασίες για την διατήρησή τους θα πρέπει να είναι όσο δυνατό πιο εναρμονισμένες έτσι ώστε να μην επηρεάζεται η εσωτερική αγορά και ταυτόχρονα να γίνονται ε, σεβαστά τα, σε, σε, σε, να γίνονται σεβαστές οι εθνικέ διατάξεις. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να διαθέτουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα προστασία δεδομένων για όλα αυτά. Μόνο δύο κράτη-μέλη δεν έχουν μεταγράψει την οδηγία αυτή τη στιγμή. Στην αξιολόγηση της, του περασμένου έτου ε, που έκανε η Κομισιόν ε, παρουσιάστηκαν ε, οι απόψει τη Europol και των κρατών μελών. Ε, και εξακολουθούν να πιέζουμε τα κράτη-μέλη να δίδουν αξιόπιστα και συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία ε, και περιπτωσιολογικές μελέτες. Ε, και έχουμε λάβει πολλές πληροφορίες. Οι αστυνομικές αρχές και οι δικαστικές αρχές στα κράτη-μέλη υπογραμμίζουν επανειλημμένα το ότι θέλουν τα δεδομένα αυτά να, είναι, να διατίθενται, να είναι διαθέσιμα αν τα χρειαστούν. Όμως, ε, πολλοί άλλοι, μεταξύ αυτών και πολλοί από εσά, εκπρόσωποι της κοινωνίας προστασία δεδομένων, ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, κάποιες επαγγελματικέ ομάδες όπως οι δικηγόροι και οι, δημοσιογράφοι ε, και οι κομισιόν, πιστεύουμε ότι η διατήρηση των δεδομένων επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ιδιωτική σφαίρα και τα, και δικαιώματα περί των προσωπικών δεδομένων. Οι οποιασδήποτε αδυναμίες θα πρέπει να βελτιωθούν. Όλα αυτά εξετάζονται στην ε, έκθεση αξιολόγησης ε, και επίσης εξετάστηκαν και στην διαβούλευση. Ε, για παράδειγμα, πιο μειωμένη και πιο αναρρωμένη περίοδος διατήρησης, ένα πολύ ε, σαφές πεδίο ε, εφαρμογής ε, και ε, συγκεκριμένος περιορισμός για το πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα. Επίσης, ελάχιστες προδιαγραφές για την πρόσβαση στα αυτά τα δεδομένα, σαφείς κανόνες για το ποιος είναι υπόλογος σε ποιον και σίγουρα χρειαζόμαστε γενικότερα μια πιο ισχυρή προστασία και πιο συνεπή προστασία. Επίσης, χρειάζεται να είμαστε λογικά συνεπείς ανάμεσα στις υποχρεώσεις για την διατήρηση των δεδομένων σε αυτή την οδηγία και στην δυνατότητα που έχουν τα κράτη-μέλη σήμερα να επιτρέπουν να διατηρούν δεδομένα σύμφωνα δυνάμει της οδηγίας ε, ηλεκτρονικής, ηλεκτρονικού απορρίτου. Ε, θα πρέπει επίσης να αποφύγουμε να χρησιμοποιούνται τα, τη, η δυνατότητα, να αποφύγουμε την δυνατότητα των κρατών μελών να χρησιμοποιούν τα στοιχεία αυτά ε, για άλλους σκοπούς εκτός αυτών που προβλέπει η οδηγία αυτή και αυτή τη στιγμή γίνεται αυτό. Ε, θα πρέπει λοιπόν να ε, εφαρμόσουμε ένα γενικότερο πλαίσιο. Ε, θα η μελλοντική αναθεώρηση τη ε, οδηγία για την ηλεκτρονική ε, προστασία δεδομένων ε, θα υποβληθεί μαζί με τι νέε μα προτάσει για την οδηγία διατήρηση των δεδομένων. Δεν μπορώ να σα δώσω συγκεκριμένη, συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα σήμερα, αλλά να σα πω ότι ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξή σας και περιμένουμε και τη δική σας νόμη. Είναι πολύ επικοδομητικά όλα όσα έχετε εκφράσει ως τώρα. Ευχαριστώ. Thank you very much, Madam Commissioner. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Θα ξεκινήσουμε με τους αγορητές των ομάδων. Για το ΕΛΚ, ο κ. Ντίας Τεμέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε. Ε, δεν αγνοούμε ότι η προστασία των δεδομένων είναι θεμελιώδες δικαίωμα που προβλέπεται από το άρθρο 8 της ε, Χάρτας των θεμελιών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο άρθρο 16 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ε, ισχύουσα οδηγία γεννήθηκε προκειμένου να εναρμονιστούν οι διατάξεις των κρατών μελών οι σχετικές με την διατήρηση των δεδομένων προκειμένου να εγγυόμαστε την διαθεσιμότητά τους για λόγους διώξεων και εκδίκασης συγκεκριμένων Όπω όπως η τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα. Όλα αυτά είναι απαραίτητα διότι ο κατακαιρματισμός σε εθνικούς ε, κανόνες ε, ε, παρεμποδίζει την δράση των δικαστικών και αστυνομικών αρχών. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε τη συνέχεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση της διατήρησης και των, των στοιχείων των ε, Ένα παράδειγμα για το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα ήταν η σύλληψη στις 4 Οκτωβρίου στην Ισπανία ενός νέου που προσπάθησε ε, να επαναλάβει την σφαγή τη Κολουμπάιν ε, στις νήσου. νήσους. Μέσω της δεδομένων που έλαβαν από την παρακολούθηση των, ε, της ηλεκτρονικής του επικοινωνίας ε, τον εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές και αποφύγαμε μια καταστροφή. Ε, ζητώ λοιπόν από την ε, Επιτροπή να προτείνει ε, ε, ταχύτατα την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου που ισχύει αυτή τη στιγμή για, το, για την διατήρηση των δεδομένων διότι εξαιτία της σημασίας και της ευαισθησίας του δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ε, ε, εφαρμόζουμε μια οδηγία που έχει τεχνικές αδυναμίες ε, που πολλές φορές παρεμβαίνει με τρόπο πολύ ομό στο δικαίωμα απορρίτου και προσωπικής σφαίρας. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά ο κύριος Λόπες Ακυλάρ για το S&D. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, είμαι μεταξύ των υπογραφώντων ε, αυτής της πρότασης. Συνεπώς συμφωνώ ε, απόλυτα με αυτούς που έλαβαν το λόγο πριν από εσά. Διότι οι ανησυχίε είναι βάσιμες. Η οδηγία αυτή ε, δικαιολογήθηκε παρουσιάστηκε μάλλον ως συνεισφορά στην καταπολέμηση εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος και ιδιαίτερως εναντίον της τρομοκρατίας. Αλλά ε, οι απόπειρε και οι ενέργειε του 2004 και του 2005 στην Ισπανία και στο, στη Μαδρίτη μάλλον και στο Λονδίνο ε, δείχνουν ότι ε, τα δικαστήρια και πολλά συνταγματικά δικαστήρια μεταξύ αυτών δίνουν, αμφισβητούν την το ότι αυτή η οδηγία, η μεταγραφή τη ε, τηρεί συγκεκριμένε αρχέ, όπω η αναλογικότητα για παράδειγμα ε, που ε, προβλέπονται από το άρθρο 8 του ε, χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το άρθρο 16 της Συνθήκης λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει στην αναθεώρηση τη οδηγίας να είμαστε πιο πετυχημένοι και να λάβουμε υπόψη τι ανησυχίε που υπάρχουν. Αυτή η πρωτοβουλία της οποίας δεν μας διευκρινίσατε το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει ε, να είναι κατά το δυνατόν λιγότερο παρεμβατική σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και να εγγυάται ε, τις αρχές, την, εφαρμή των αρχών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια η κυρία Ιντβέλτ από τους Φιλελεύθερους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, συνάδελφοι, αυτή η οδηγία ε, ήταν κάτι ασφαλμένο ευθύ εξ αρχής. Ας δούμε τι έγινε κατά το παρελθόν. Ο λόγος για τον οποίο ψήφισε για την πρόταση για τη δεκάτη στοιχείων του Κοινοβούλιο είναι διότι δεν συμφωνούσαν τα κράτη-μέλη. Δεν υπήρχε ομοφωνία. Το θυμόσαστε. Ε, πολλά κράτη-μέλη δεν το ήθελαν. Και γι' αυτό ψηφίσαμε. Και αυτός ο λόγος. Μέχρι σήμερα ε, προσπαθούν να αποφύγουν την παρέμβαση την κοινοβουλευτική. Δεύτερον, εξυπηρετεί κάποιο σκοπό, είναι κάτι χρήσιμο. Ε, γίναμε ασφαλέστεροι μετά το 2005-2006. Παρά το γεγονός ότι η αξιολόγηση έγινε μετά από μεγάλες καθυστερήσεις, δεν υπάρχει ίχνος απόδειξης, συνάδελφοι, ίχνος λέγω απόδειξης, που να δείχνει ότι συμβάλλει στην ασφάλειά μας. Όλες οι δηλώσεις περί αναγκαιότητας της οδηγίας ε, δράζονται επί υποθέσεων και σε τίποτα άλλο. Ακόμα δεν έχουμε δυστυχία. Εξυπηρέτησε τον σκοπό της εναρμόνισης. Νομίζω ότι τον έφεραν συνάδελφοι. Δεν έχει καταφέρει κάτι τέτοιο. Δεν το έχει καταφέρει. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός ευθύς εξ αρχής. Άλλωστε, διότι τα κράτη-μέλη επέλεξαν να αποζημιώσουν ε, τις εταιρείες για το κόστος. Θεωρήθηκε παραβίαση των συνταγμάτων διαφόρων χωρών. Μπορείτε να πείτε συνάδελφε ότι είναι τεχνικό θέμα αυτό. Ότι εφαρμοστικός νόμος θεωρήθηκε αντισυνταγματικός. Αλλά φαίνεται να είναι αδύνατο να βρεθεί ένας τρόπος να εφαρμοστεί με έναν τρόπο που να ταιριάζει με το Σύνταγμα. Στη χώρα μου, μια έκθεση έδειξε ότι υπάρχει ευρεία κατάχρηση. Τα στοιχεία κρατούνται επί πολύ μεγαλύτερο χρόνο από πολλούς περισσότερους από ό,τι επιτρέπεται. Κάνει κανείς κάτι? Όχι. Έχουμε λοιπόν ένα νόμο που ψηφίστηκε, που δεν εξυπηρετεί κάποιο σκοπό, φαίνεται να παραβιάζει το Σύνταγμα, ε, γίνεται ευρέω κατάχρηση και βεβαίω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη λένε υπέροχο νόμο, θέλουμε περισσότερου σαν κι αυτού. Επίτροπε, δεν πρέπει να περιμένουμε μέχρι να γίνει αναθεώρηση. Θα πρέπει να ανακληθεί σήμερα η ισχύ αυτού του μέτρου. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος είναι ο κύριος Άλμπρεχτ που έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Μιλούμε για διακράτηση των δεδομένων πλαισίου των τηλεπικοινωνιών και των 500 εκατομμυρίων πολιτών ανα πάσα στιγμή. Όχι σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, όχι όταν θεωρούνται ύποπτοι, αλλά ανα πάσα στιγμή διαρκής παρακολούθηση κάθε ενός πολίτη. Αντιλαμβάνεστε περί τι σοβαρής ε, παραβίασης των προσωπικών δεδομένων και των θεμελιωδών ελευθεριών αυτών των ανθρώπων μιλάμε. Και διερωτώ εάν οι προλαλήσαντες όπως και οι προλαλήσαντες, εάν έχουμε αποδείξει, αν μπορούμε να αποδείξουμε ότι αυτή η οδηγία, αν αυτή η διακράτηση των προσωπικών δεδομένων είναι είτε απαραίτητη είτε επαρκής ώστε να ε, βοηθήσει στην δίωξη εγκλημάτων μέσα από το διαδίκτυο, επί παραδείγματι. Δεν έχω δει πουθενά τέτοια απόδειξη και αν αντιληφθούμε πόσο σοβαρά είναι τα προβλήματα και πόσο σημαντική η ανάγκη να καταπολεμηθεί η εγκληματικότητα, κυρίως μέσα από το διαδίκτυο, χωρίς όμως να έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει αδίποτε αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της, ε, μεταξύ της διακράτησης των προσωπικών δεδομένων αυτών και της καταπολέμησης των διαδικτυακών εγκλημάτων, είτε πρόκειται για κράτος που έχει εισαγάγει την νομοθεσία και την εφαρμόζεται μη. Βλέπουμε ότι πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο είναι ακριβό, πρόκειται για χρήματα λέει, τα οποία μας λείπουν από αλλού, όταν έχουμε ε, παραδείγματι την αδυναμία σε ένα αστυνομικό τμήμα να εξασφαλίσουμε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ε, νομίζω ότι η κατάσταση είναι μάλλον ανησυχητική και πρέπει να μας βάλει στις σκέψεις. Ευχαριστώ Σας ευχαριστώ πολύ. πολύ. Η κυρία Ένς στην επόμενη. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θέλω να πω ότι δεν επιλύει προβλήματα. Είναι πρόβλημα η διακράτηση προσωπικών δεδομένων και επιτρέψτε μου ως προς τη χρησιμότητα να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πρόσφατα είχα πάει στη Δρέσδη όπου είδα μία περίπτωση να, να χτυπάει κάποιος ε, την πόρτα μιας ε, γριάς ε, κυρίας για να, να χτυπάνε στην αστυνομία την πόρτα μιας γριάς κυρίας για να ε, ψάξουν κάποια στοιχεία της. Διερωτώ με αν με αυτόν τον τρόπο θέλετε ότι μπορείτε να αντιμετωπίσετε την εγκληματικότητα. Πρότεινα, λοιπόν, θα πρότεινα λοιπόν κυρία Μάλστρομ να απευθύνεται στους υπουργούς των εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την εξής πρόταση. Αντί να καταργούν θέσεις αστυνομικών και δικαστικών υπαλλήλων και προσωπικού στις χώρες τους να ενισχύσουν τα σχολεία, τις σχολές αστυνομικών, τις σχολές δικαστών, να βελτιώσουν την κατάρτισή τους ώστε να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους προς όφελος των πάντων, της κοινωνίας και κυρίως των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Πάσκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο, κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Κατά την, ιδέα, κατά την άποψη του αρμοδίου την προστασία των, δεδομένων στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα την άποψη των αρμοδίων φορέων ε, στη Γερμανία, τη Ρουμανία και Πολωνία η οδηγία αυτή που επιτρέπει στις εταιρείε τηλεφώνων να κρατήσουν στοιχεία για τους διάφορους χρήστες αποδέκτη τηλεφωνήματο, εκείνο που κάνει το τηλεφώνημα κλπ. για έρευνε εγκλημάτων για έξι μήνε μέχρι και δύο χρόνια δεν είναι κάτι που ταιριάζει με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη δυτική ζωή. Λοιπόν, κυρία Επίτροπε, θα πρέπει να πάρουμε υπεύθυνη απόφαση. Είτε να ακυρώσουμε αυτή την απόφαση και να αφήσουμε τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν πώ θα αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα ή αν υπάρξει συμφωνία ε, για δικαστική συνεργασία και αστυνομική συνεργασία σε ποινικέ υποθέσει, να γίνεται κάτι τέτοιο, τότε χρειαζόμαστε κοινού ευρωπαϊκού ε, νόμου. Χρειαζόμαστε νέα νομοθεσία που να αντιστοιχεί όμω στην νοοτροπία που ακολουθεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και έρχεται αρκετό χρόνο να πάρετε υπεύθυνε απόφασει προ αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριο ε, Κοέλιο. Κυρίε και κύριοι, Κύριε Επιτροπέ, ο κύριος Δεμερά μας υπενθύμησε τις ε, ε, συνθήκες ε, που επικράτουσαν κατά την υιοθέτηση αυτής της οδηγίας. Είναι προφανές ότι τα κράτη-μέλη επωφελήθηκαν ιδιαίτερως από την προθεσμία που ορίζεται για την διατήρηση των δεδομένων. Ε, αυτοί οι 24 μήνες ε, είναι ένα από τα εργαλεία πιο πολύ χρησιμοποίησαν τα κράτη-μέλη. Διάφοροι ομιλητέ αναφέρθηκαν στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με την ε, μεταγραφή στο εθνικό δίκαιο με διαφορετικό τρόπο. Σχεδόν όλοι οι ομιλητέ υπογράμμισαν σωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σχετικά με την προστασία των θεομελιών δικαιωμάτων και του δικαιώματο προστασίας προσωπική ζωή. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Εγώ είμαι μεταξύ αυτών που, ε, ε, ε που τους άρεσαν οι απαντήσει της κυρίας Μάλστρομ. Η κυρία Μάλστρομ αντιλαμβάνεται τα προβλήματα τη οδηγία, όπως για παράδειγμα ότι πρέπει να περιοριστούν οι περίοδοι διατήρηση, να οριστεί καλύτερα το πεδίο εφαρμογή κλπ. Όλα όσα είπε η κυρία Μάλστρομ αποτελούν τμήμα της ε, προσπάθειας αναθεώρησης αυτή τη οδηγία. προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί. Αυτό που με ανησυχεί όμως είναι το χρονοδιάγραμμα, ο χρόνος. Εγώ ήμουν σίγουρος ότι μέχρι το τέλος του χρόνου η Κομισιόν θα μας υπέβαλε μια καινούργια πρωτοβουλία. Η κυρία Μάλστρομ είπε ότι αυτό σίγουρα δεν θα γίνει μέχρι το τέλο του χρόνου, αλλά δεν μα δίνει και ε, χρονικό ορίζοντα. Ε, οπότε τι σημαίνει αυτό, ότι σε έξι μήνες, ένα χρόνο και δύο χρόνια από σήμερα πάλι θα ρωτάμε την Επίτροπο πότε θα υποβάλει την αθεώρηση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δρούτσας, ο κύριος Δημήτρης Δρούτσας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε και εγώ ενώνω τη φωνή μου με τις διαμαρτυρίες και που ακούστηκαν στους συναδέλφους και τα επιχειρήματα που έβαλαν συνάδελφοι που, μίλησαν προηγουμένως. Δεν θέλω να επαναλάβω, δεν χρειάζεται τα ήδη υποθέντα αλλά θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα του πότε θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρότασή της. Δεν ξέρω αν σας αντελήφθη ορθώς. Είπατε ότι δεν προτίθεστε να υποβάλλετε την πρότασή σας φέτος. Και ρωτώ, πότε του χρόνου. Έχουμε 12 μήνες μπροστά μας. 12 ε, μήνες έχει ο επόμενος χρόνος. Μπορείτε να ξεκαθαρίσετε πότε. Μέσα στον επόμενο χρόνο. Πότε θα υποβάλλετε την πρόταση. Το λέω αυτό διότι θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι τώρα ασχολούμεθα με το πακέτο μεταρρύθμισης των προσωπικών στοιχείων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί το θέμα αυτό ότι έχει πραγματική προτεραιότητα και έχει αφοσιωθεί στις προσπάθειες και για τον προτινόμενο κανονισμό και την οδηγία. Και θα πρέπει να εναρμονίσουμε και την ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σχετικά με αυτό το θέμα. Και θα πρέπει να ήρθε και ο καιρός για την οδηγία για την ηλεκτρονική προστασία ιδιωτικής ζωής. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είναι πιο δυναμική έναντι των κρατών μέλων. Ακόμα και αν πρόκειται για τα ούτως αποκαλούμενα ευαίσθητα θέματα για τα κράτη-μέλη. Και θα ήθελα να πω, Επίτροπε, κλείνοντα, ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα θα βρίσκεται έναν ενθουσιώδη σύμμαχο στις προσπάθειες που καταβάλλετε για τη μεγαλύτερη προστασία των προσωπικών στοιχείων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και μπορείτε πάντα να βασίζεστε στην πλήρη συνεργασία μαζί μας, στην πλήρη στήριξή μας. Όμως, ταυτόχρονα, να τονίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα θα είναι έτοιμο να πολεμήσει και να υπερασπιστεί για τις αρχές, να υπερασπιστεί τις αρχές του θα είναι υπέρ τη προστασία των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών, κυρίω όταν πρόκειται περί θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Επόμενο είναι ο κ. Σλίτα. Ε, eh, ευχαριστώ. Ε, σίγουρα χρειαζόμαστε μια πιο αναλογική οδηγία. Αλλά τι σημαίνει αναλογικότητα. Αναλογικότητα για κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία, για κάθε πολίτη. Ε, Κανένα δεν θα πρέπει να διαφεύγει δηλαδή από αυτήν την οδηγία. Ακόμα και ο George Orwell ε, δεν είχε φανταστεί ένα τέτοιο φιάλτη. Και ο George Bush δεν είχε καν προτείνει κάτι τέτοιο. Ε, κινούμαστε στα όρια της παράνοιας. Ε, τι θα πρέπει να κάνουμε. Ε, ε, είναι σαν να ψάχνουμε μια καρφίτσα μέσα σε ένα δεμάτι με άχυρα. Ε, είναι δυνατόν ε, να μας τσιμπήσει, υπάρχει τέτοια περίπτωση, ε, αυτή την οδηγία έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι αναλογική, προφανώς, δεν είναι αποτελεσματική. Θα πρέπει να την αποσύρουμε το συντομότερο δυνατό. Να... Δεν χρειάζονται μελέτες για να αποδειχθεί αυτό. Δεν υπάρχουν ε, ενδείξαν ότι είναι ε, αποτελεσματική. Κύριε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, πριν να διατυπώσω την ερώτησή μου, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι πριν από μια εβδομάδα το Πολωνικό Κοινοβούλιο υιοθέτησε νόμο για τις τηλεπικοινωνίες, όπως περίμενε από καιρό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με πρόνοιες για όρια προθεσμίες δηλαδή ε, πιο σύντομες διακράτησης των στοιχείων. Η Πολωνία δηλαδή τώρα πια είναι και αυτή χώρα με διατάξεις σύμφωνες με το ευρωπαϊκό δίκαιο και επεξεργαζόμαστε νέες προτάσεις για την διακράτηση στοιχείων και την πρόσβαση σε αυτά. Θα θέλαμε ως εκ τούτου να γνωρίζουμε τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι προτάσεις σκοπεύει να καταθέσει ώστε την νομοθεσία μας να την προσαρμόσουμε αναλόγως. Και είναι πολλές οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις οι οποίες έχουν μελετήσει το θέμα αυτό, έχουν ασκήσει πίεση στις αρχές, διότι θεωρούν ότι αυτές ε, οι διατάξεις παρεμβαίνουν, παραβιάζουν τις της ελευθερίας των πολιτών και νομίζω ότι θα πρέπει να ακούμε όχι μόνο τους πολίτες αλλά και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις οι οποίες ε, υπογραμμίζουν ιδιαίτερα τη σημασία του ιδιωτικού βίου. Ερωτώ λοιπόν εάν έχει μελέτες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς τι συνέπειες μπορεί να έχει η περιστολή της περίοδου διακράτησης ως προς την αποτελεσματικότητα της ε, επιβολής του νόμου, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση των σοβαρών εγκλημάτων, τα χειρή επιχειρήματα δηλαδή που χρησιμοποιείτε όταν μιλάτε για την ανάγκη διακράτησης. Αλλά θέλω συγκεκριμένα στοιχεία. Έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματική αυτή η μέθοδος, ιδιαίτερα στα θέματα της παιδικής πορνογραφίας. Βοηθάει καθόλου στην καταπολέμηση των εγκληματιών. Ευχαριστώ και για ένα λεπτό τώρα η κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ. Έχουν ε, καλυφθεί σχεδόν όλα τα επιχείρηματα, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω ουσιαστικά γιατί θέλουμε να έχουμε αποθηκευμένα στοιχεία. Αποθήκευση. Τι σημαίνει, αν αποθηκεύσω τρόφιμα στην αποθήκη μου, κάποια στιγμή πρέπει να τα χρησιμοποιήσω, κάποιο στόχο έχουν, πρέπει να καταναλωθούν. Άρα και τα δεδομένα που θα αποθηκεύουμε θα πρέπει να αξιοποιούνται για να καταπολεμήσουν σοβαρά εγκλήματα, τρομοκρατία κτλ αλλά ίσως και για μικρότερης βαρύτητας αδικήματα και έτσι αρχίζει η διακράτηση δεδομένων ε, που αρχικά δεν είχαν υπολογιστεί ότι θα διακρατούνται. Άρα λοιπόν και ο όγκος των δεδομένων θα πρέπει να αξιολογηθεί μαζί με τη σκοπιμότητα της διακράτησής τους, μαζί με την ενδεχόμενη κατάχρηση αυτών. Είναι πολλές οι πρακτικές που πρέπει να αναθεωρηθούν, δεν πρέπει να μας σταματά κανένα ταμπού προς την αμφισβήτηση των, της χρήσης αυτών των δεδομένων και πάση περιπτώσει κύρια αρχή πρέπει πάντοτε να είναι η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και σε περίπτωση αμφιβολίας ακόμη να προχωρήσουμε και στην κατάργηση της οδηγίας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ρωμέρο Λόπες, τελευταία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Μάλστρομ, όταν μιλάτε για την αναθεώρηση, ε, είπατε ότι θα γίνει μέσα στο πλαίσιο της αρχής αναλογικότητας. Ε, Όλες οι οδηγίες λένε ότι βρίσκονται στα όρια της αναλογικότητας. Αυτό το λένε όλες οι οδηγίες. Ε, και με, την, ε, και τα, με τα Μητρό Επιβατών και, και με όλες τις άλλες οδηγίες. Το πρόβλημα είναι ότι όταν έχουμε μια οδηγία για, ε, η οποία ε, αφορά ειδικέ περιπτώσεις για τις οποίες είναι δυνατόν να γίνει παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πολύ δύσκολο πλέον το καθήκον μας διότι ποια είναι αυτά τα σοβαρά αδικήματα γιατί οκτώ χώρες δεν μιλούν για σοβαρά αδικήματα μιλούν για οποιοδήποτε τύπου αδίκημα στη μεταγραφή ε, είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστούμε τον αγώνα κατά της κατά των, των αδικημάτων ε, διότι ε, σπανίως ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Ε, θα πρέπει πραγματικά να περιορίσουμε πάρα πολύ το πεδίο εφαρμογής. Δεν είναι δυνατόν να αφήνουμε ανοιχτό το παράθυρο για τέτοιου είδους υπερβολές. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε τη διαδικασία προσέξης προσοχής του Προέδρου. Κατστιάε. Η κυρία Μπασέσκου είναι η πρώτη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η εφαρμογή τη οδηγία και ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο ήταν πρόκληση για πολλά κράτη-μέλη και υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία δεν την έχουν ενσωματώσει στη δική του ανενομή τάξη. Οι, οι λόγοι σχετίζονται με το επίμαχο θέμα τη παραβίαση τη προστασία τη ζωή. Η ίδια κατάσταση ήταν και στη Ρουμανία. Το νομοσχέδιο θεωρήθηκε αρχικά ε, αντισυνταγματικό. Μόλις φέτος ενσωματώθηκε στην νομοθεσία μας η οδηγία. Ε, γι' αυτό πιστεύω ότι ένα νέο πλαίσιο θα πρέπει να αναπτυχθεί ούτως ώστε να καταργηθούν αυτά τα επίμαχα ζητήματα. Θα πρέπει να λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα συντάγματα των κρατών μελών όταν ετοιμάζει προτάσεις. Οι προτάσεις επίσης θα πρέπει να διαφυλάσσουν το δικαίωμα τη προστασία της ιδιωτικής ζωής. Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή τη να τροποποιήσει την οδηγία πέρσι, δεν το έκανε μέχρι τώρα. Κατά την άποψή μου, η νέα πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι το τέλο του έτου, ούτω ώστε να αποφευχθούν προβλήματα και σε άλλα κράτη-μέλη. Να μην προσφύγουν άλλα κράτη-μέλη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο. Η κυρία Τσικάου είναι η επόμενη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κυρία Επίτροπε τον Ιούνιο του 2011 είπε, έστειλα γραπτή ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ρωτούσα κατά πόσο θεωρούσε ότι η αναθεώρηση της οδηγίας ε, για την διακράτηση στοιχείων θα λάμβανε χώρα, ούτως ώστε να υπάρχουν συνεπείς νόμοι και διατάξει για τη διακάτηση στοιχείων σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών μελών, τα συντάγματα των κρατών μελών και σύμφωνα με, τις, ε, με την ε, Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, ώστε να μην παραβιάζεται το δικαίωμα προστασία ελεύθερη διακίνηση ελεύθερης μετακίνηση και προστασία ε, της ιδιωτικής ζωής. Στις 12 ε, Αυγούστου του 2011 στείλατε απάντηση και εκεί αναφερθήκατε σε διαβουλεύσεις που είχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης, με την κοινωνία των πολιτών, με τα κράτη-μέλη, με τους εκπροσώπους ε, του τομέα και τις δικαστικές αρχές. Ε, είπατε ότι είχατε σημειώσει ε, τις διάφορες απόψεις σχετικά με ενδεχόμενες λύσεις και ότι επρόκειτο να προβείτε σε μια αξιολόγηση των λύσεων μέσα σε μια έκθεση αξιολόγησης. Αυτή η έκθεση αξιολόγηση ποιον, είναι έτοιμη, θα δημοσιευτεί και αν δημοσιευτεί πότε. Ευχαριστώ. Η κυρία Λίχτενμπεργκερ είναι η επόμενη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Είμαι απογοητευμένη διότι δεν δώσατε για άλλη μια φορά ε, συγκεκριμένες ε, οι πληροφορίες για το πότε σκοπεύετε να καταθέσετε τη νέα πρόταση. Μας ε, λέγεται πάντως ότι δεν ε, θα διδόταν η ίδια λύση, νομοθετική λύση για τα προσωπικά δεδομένα και τη διακράτησή τους σήμερα. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό για μένα. Είναι πολύ ενισχυτικές όλες οι αναφορές ε, ως προς την χρήση, την εφαρμογή του συστήματος. Είναι πολλές οι παραβιάσεις και μπορεί να είχε προβλεφθεί για εφέτος ένα, ε, αλλά δεν βλέπουμε ουσιαστική απόδοση αποτελέσματος από την νομοθεσία και λόγω της μη εφαρμογής από ορισμένα κράτη-μέλη, αλλά και πάνω απ' όλα γιατί είναι ανοιχτή η νομοθεσία αυτή σε κάθε τύπου καταστρατήγηση. Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κρυθεί και από αυτό το ζήτημα, κύριε Επίτροπε. Παρακαλώ, επιτέλους, καταθέστε αυτή την πρόταση τροποποίηση της νομοθεσίας. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Έγκστρομ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Επίτροπε, πρόκειται για μια οδηγία αποτυχημένη που επηρέασε αρνητικά την προσωπική ζωή των πολιτών μας. Δεν έχει τίποτα το θετικό, δεν, έχει, δεν υπάρχει τίποτα που να δείχνει την αποτελεσματικότητά της στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Η οδηγία αναφέρει ότι η Κομισιόν θα αξιολογήσει ε, την εφαρμογή της ε, μέχρι το Σεπτέμβριο του 2010. Δεν έγινε τίποτα τέτοιο. Ε, Μα αναφέρονται κάποιες ιστορίες, ε, θεωρητικές πιο πολύ, το για το κατά πόσον ε, η διατήρηση των δεδομένων μπορεί να βοηθήσει. Αλλά όλα αυτά είναι πιο πολύ θεωρητικά. Πώς είναι δυνατόν η Κομισιό να επιβάλλει κυρώσει στη Σουηδία γιατί δεν έχει μεταγράψει αυτήν την οδηγία, ενώ ε, δεν υποβάλλει την αξιολόγηση η οποία προβλεπόταν από την οδηγία. Um, Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και συνάδελφοι. Η διακράτηση στοιχείων και τα σχετικά μέτρα που λαμβάνονται οδηγούν σε ευαίσθητα προβλήματα όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα κλπ. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής διακινδυνεύει λόγω της χρήσης των στοιχείων. Κυρίως άμα υπάρχει ένα οριζόντιο μέσο για την χρήση των στοιχείων που διαβάζονται μέσω επικοινωνίων. Με τον κόσμο μετά την 11η Σεπτεμβρίου οι διάφοροι νομοθέτε δεχόταν τρομερέ πιέσει να δείξουν αποφασιστικότητα και ισχύ στην καταπολέμηση τη διεθνού τρομοκρατία και του οργανωμένου εγκλήματο. Σφάλματα και καταχρήσει έγιναν πάρα πολλά. Αλλά οι συζητήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον καλύτερο τρόπο να αντιμετωπιστεί το σοβαρό έγκλημα ωφελήθηκαν γιατί το περιβάλλον ήταν πολύ πιο ήρεμο, κυρίως σε συγκρίση με τι ΗΠΑ. Η Ευρώπη δεν αμέλησε τι ευθύνε που έχει στον τομέα αυτόν. Ούτε θα πρέπει να μην αξιολογήσει την αναλογικότητα και την αποτελεσματικότητα ή ονδήποτε μέτρων ε, ασφαλείας που ανταποκρίνονται σοβαρές απειλές. Ε, οι ζωές απειλούνται. Ε, το ταχύτερο δυνατόν θα πρέπει να κάνει αναθέω Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο πιο γρήγορα το επιτρέψει η ολοκλήρωση τη αξιολόγηση συνεπιών. Ευχαριστώ, Λε Πρόεδρο, για τα τελικά σχόλιά τη. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Επίτροπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσήλωσή σας. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα, αλλά Παρακαλώ αντιληφθείτε ότι η διατήρηση των στοιχείων θα παραμείνει γιατί την υποστηρίζουν τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη δεν πρόκειται να δεχτούν προτάσεις κατάρρισής της. Το πρόβλημα είναι απλώ ότι υπάρχουν 27 διαφορετικέ ε, εκδοχέ τη διατήρηση. Δεν έχουμε κοινού κανόνε. Αυτό θα πρέπει να επιλύσουμε. Ε, κάναμε την αξιολόγηση τον Απρίλιο του 2011. Είχαμε ε, ε, στοιχεία ε, περιπτωσιολογικά, αυτό είναι αλήθεια, αλλά έχουμε μαζέψει πάρα πολλές πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιήθηκε η διατήρηση δεδομένων στην καταπολέμηση του εγκλήματος, στην εξάρθρωση ε, συμμοριών, ε, στην συλλογή στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν από τους αγγελείς. Μπορώ να σας ενημερώσω για αυτά. Ξανά, το έχουμε ξανακάνει άλλη μια φορά. Μπορώ να, το, να σας ξαναενημερώσω λεπτομέρως για όλες αυτές τις περιπτώσεις. Καταλαβαίνω βέβαια τις επικρίσεις. Ε, και συμφωνώ με πολλά από αυτά, αλλά δεν παρακολουθούνται 500 εκατομμύρια άτομα ε, κατά σύστημα. Ε, τα, πρόκειται για στοιχεία τα οποία διατηρούν εμπορικές επιχειρήσεις και μπορούν να τα... να, έχουν πρόσβαση σε αυτά αστυνομικέ και δικαστικές αρχές υπό συγκεκριμένες συνθήκες και όρους υπάρχει δικαστικός και δημοκρατικός έλεγχος στα κράτη-μέλη. Τώρα, υπάρχουν βέβαια προβλήματα και αδυναμίε με την οδηγία. Αυτά τα υπογράμισε η μελέτη αξιολόγηση και αναφέρθηκα και εγώ σε αυτά προηγουμένως. Δεν έχει εξασφαλιστεί επαρκής εναρμόνιση και ε, ε, δεν έχει ξεκαθαριστεί ποιος έχει πρόσβαση, ε, πώς προστατεύονται και για ποια περίοδο διατηρούνται. Θα πρέπει να τα ενοποιήσουμε και να βραχύνουμε την περίοδο διατήρησής τους. Επίσης πρέπει να δούμε πώς επηρεάζει η οδηγία αυτή την προσωπική ζωή και το απόρριτο τη προσωπική ζωή. Όμω είναι σημαντική η διατήρηση των δεδομένων. Χρειαζόμαστε ένα ε, ευρωπαϊκό πλαίσιο και γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό μαζί να προσπαθήσουμε να το λύσουμε μαζί με πολλά άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, υπάρχουν κάποια ε, κενά και παραθυράκια στην οδηγία ε, της ηλεκτρονικής ιδιωτικής ζωής. Το, είδα, το είπατε και εσείς αυτό. Και οι αναθεωρήσεις των δύο οδηγιών θα πρέπει να πάνε παράλληλα, μαζί, ταυτόχρονα. Γι' αυτό το λόγο και δεν μπορώ να σας δώσω και συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα για το πότε θα γίνουν όλα αυτά. Αλλά ο στόχος είναι να διαθέτουμε μια στέρεη βάση για την προστασία των δεδομένων και θέλω να συνεργαστώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαδικαστικό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση σχετικά με, με τους κανόνες που ισχύουν. Αν θέτουμε ερώτημα προς την Επίτροπο, θα θέλαμε να ακούσουμε απάντηση. Και ένα ερώτημα δεν το απάντησε μέχρι τώρα η Επίτροπος. Το εξή. Αν το πάγωμα των στοιχείων, όπως γίνεται στις ΗΠΑ, αν αξιολογήθηκε σωστά, διότι από τα στοιχεία δεν είναι σαφές. Αν έχεις ένα δίκτυο ε, εμπόρων ναρκωτικών. Υπάρχουν υπόνοιες επιμακρών γι' αυτό, είναι σαφέ. Και ένα πάγωμα στοιχείων για κάθε άτομο θα λειτουργούσε εξίσου καλά, διακόπτει ο πρόεδρο. Είπατε ότι είναι διαδικαστικό. Κύριε Επίτροπε, ίσω αν μπορούσατε να απαντήσετε. Ε, συγγνώμη, έπρεπε να το είχα αναφέρει. Το quick freeze, το πάγωμα για σύντομο χρονικό διάστημα, είναι κάτι διαφορετικό από τη διατήρηση των στοιχείων και το εξετάζουμε δεν θεωρείται σαν εναλλακτική για τα κράτη-μέλη όσον αφορά τη διατήρηση των στοιχείων. Κάνουμε μελέτη και για αυτό που είπατε και θα το παρουσιάσουμε μέσα στο γενικότερο πλαίσιο και στη συγκεκριμένη πρόταση. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, λέει Πρόεδρος. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Το επόμενο σημείο που έχουμε στην τη διάταξη είναι η δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, με την Ιαπωνία για εμπορικά θέματα. Α, θα ήθελα να δώσω καταρχάς το λόγο.